Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με αυτό που έπρεπε να ξεκινήσει το πρωί, τις ανακοινώσεις της Προέδρου, αλλά είχαμε δουλειές. Γιατί είχατε αργήσει κιόλας. Να σας υπενθυμίσω πως ακυρώνεται η συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας και ανταυτού έχουμε Δευτέρα 6.30 με 9.30 ακρόαση Νίμιτσα, ακρόαση του κυρίου Στυλιανίδη, τρίτη 6 με 9. Και επίσης θα κάνουμε και μία ερώτηση στη κυρία Μάνστρομ ε, και στην ακρόαση Μοργερίνη στις 6.30. Από μία ερώτηση σε αυτές τις ακροάσεις. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε ακρόαση. Μόλις μάθαμε, μόλις μου δώσαν εμένα από τη άσκηψη των Προέδρων ένα σημείωμα για το χρόνο ομιλίας. Κάθε ακρόαση θα έχει 25 ερωτήσεις, 11 ΕΛΚ, 10 σοσιαλιστές, ECR 5, φιλελεύθεροι 5, γκουε 4, Πράσινη 4, EFTD 4 και μη εγγεγραμμένοι 2. Αλλά θα τα λάβετε αυτά και προφανώς οι πολιτικές ομάδες θα μοιράσουν το χρόνο ομιλίας. Οπότε θα τα δείτε από τους συντονιστές σας. Αυτά λοιπόν για τις ακροάσεις που είναι πολύ σημαντικές. Ακυρώθηκε λοιπόν η συνεδρίαση της επόμενης ε, εβδομάδας. Αλλά σήμερα στις 4.30 σε άλλη αίθουσα, όχι εδώ, 2Q2 στο δεύτερο όροφο θα έχουμε παρουσίαση των υποψηφίων 4 και 4 τις παρουσιάσεις ε, των υποψηφίων για το βραφείο Ζαχάροφ. Έχουμε προσκληθεί μαζί με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε 15 μέρες από σήμερα 5 Οκτωβρίου θα έχουμε μια ψηφοφορία το πρωί σε 7 με συγχωρείτε ψηφοφορία για το βραβείο Ζαχάροφ σημειώστε το δεν ξέρω ακριβώς την ώρα θα το κανονίσουμε αυτά με τις ανακοινώσεις της Προέδρου μετά την έμπολα που φαντάζομαι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ως ακρόαση. Βλέπουμε πως υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα απευθύνω μια επιστολή στην υπατή εκπρόσωπο για να γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν επιγόντως. Και θα στείλουμε βεβαίως το σε όλους. Δύο πράγματα λοιπόν έχουμε στην μερίσια διάταξη. Πρώτα απ' όλα συζήτηση. Τρία, με συγχωρείτε κλιματική αλλαγή και ψηφοφορία. Αλλά πριν γίνει αυτό. Ο κύριος Κρέκ Μακουέιτ, πού είναι? Από την Κομισιόν. Εδώ είστε. Α, μάλιστα. Ε, φοράω τα γελιά εδώ πέρα για το διάβασμα. Δεν σας βλέπω εκεί κάτω. Έχετε να μας πείτε τίποτα. Όχι, ωραία, ευχαριστούμε. Περνάμε λοιπόν κατευθείαν στο σημείο 7 έχω τα χαρτιά μου για την διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Να σας ενημερώσω γιατί το συζητάμε. Όπως θα ξέρουν οι συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υιοθετεί ένα ψήφισμα εν ώψη της διάσκεψης των μερών της λεγόμενης ε, που λαμβάνει χώρα τον Δεκέμβριο. Τα μέρη είναι τα μέρη που έχουν υπογράψει την ε, σύμβαση του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Η Επιτροπή αρμόδια είναι αυτή του περιβάλλοντος, αλλά πάντα και η δικιά μας η Επιτροπή ε, κάνει ένα ψήφισμα, το οποίο μπαίνει στο ψήφισμα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, μετά θα ε, ψηφίσει και το ψήφισμα μετά θα πάει στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Πρέπει λοιπόν να βιαστούμε για να πάει να μεταφραστεί, να ψηφιστεί για να ληφθεί υπόψη αρχές Νοεμβρίου στην ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος και να ψηφιστεί τον Νοέμβριο. Τα γνωρίζετε το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα το συζητήσαμε στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το οποίο λαμβάνει σήμερα χώρα στη ΣΥΠΑ όπου συγκεντρώνονται οι ηγέτες να δουν τι θα κάνουν και πώς θα προετοιμαστούν για τη διάσκεψη των μερών στη Λίμα το Δεκέμβριο και για, την, για το Παρίσι του χρόνου όπου ελπίζουμε επιτέλους μετά τις αποτυχίες της Κόπενχάγης να έχουμε μια συμφωνία παγκόσμια. Είχαμε λοιπόν την συζήτηση, λάβατε μέρος πολλοί από σας και εγώ είχα αναφέρει πως όταν είχα δει στην Κένια από πρώτο χέρι κόσμο που έχει ήδη καταστραφεί το βιός του πλέον λόγω της ξηρασίας και εκεί πέρα κατάλαβα πως συνδέεται αυτό το θέμα με την ανάπτυξη και γι' αυτό πάντα εμείς προετοιμάζουμε ένα ψήφισμα. Έχουμε λοιπόν ένα ψήφισμα, αλλά επειδή αργήσαμε να το στείλουμε για μετάφραση, δεν το έχουμε μεταφρασμένο. Δεν ξέρω αν έχετε το έγγραφο εργασίας. Μάλιστα. Οπότε εγώ είπα να σας μοιραστεί το έγγραφο εργασία. Έχει μοιραστεί με email. Τώρα σα το μοιράζουν. Έχουμε κάποια πράγματα σχέδιο ψηφίσματο που θα μεταφραστούν ε, την επόμενη εβδομάδα και μετά βεβαίω. θα έχουμε στις 3 Νοεμβρίου την ε, ψηφοφορία έχουμε μια συνεδρίαση ειδικά για αυτό το θέμα. 14 Οκτωβρίου, 12 η ώρα, προθεσμία για τροπολογίες. Έχετε λοιπόν τώρα μια ιδέα για τα βασικά του ψηφίσματος αυτού. Το βασικό είναι από τη σκοπιά της ανάπτυξης ε, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει μια αξιόπιστη πρόσφορα Δηλαδή, ε, πρώτα απ' όλα να κανονίσουμε τα του οίκου μας και μετά να έχουμε ένα πακέτο να προτείνουμε ένα στόχο για το 2030 και πολιτικές και βεβαίως ε, τι δεσμεύσεις που είχαμε κάνει το 2009 για το ε, πράσινο ταμείο να ζητήσουμε και από τους νέους επιτρόπους να κάνουν κάτι γιατί τις επόμενες εβδομάδες θα συζητήσουμε τους ε, στρατηγικούς αυτούς ε, στόχους ανάπτυξης και βεβαίω η διαδικασία στον ΟΗΕ και στο COP21 θα είναι παράλληλη. Οπότε θέλουμε ακριβώ οι επίτροποι να συνεργαστούν. Ε, ανάπτυξης, κλίματος, ε, για να δουν αυτά τα ζητήματα μαζί. Αυτές είναι οι νέες εξελίξεις. Τώρα περιμένω από εσάς ε, το τι θα γίνει Κάθριν πρώτη και μετά οι υπόλοιποι. Κοιτάξτε. Έχω την εντύπωση ότι πώς το λέμε αυτό το πράγμα, το σκεπτικό ας πούμε εκεί μπροστά πρέπει να γράψουμε κάτι παραπάνω για τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά στις αναπτυσσόμενες χώρες και την Ιρλανδία. Η κοινή συνέλευση ΑΚΕ ΕΟΚ θα γίνει τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου και την προηγούμενη φορά έγινε στη Σαμόα και μας πίεσαν πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση του επίπεδου της θάλασσας. Πρέπει κάτι να βάλουμε και εκεί. Θα μάθουμε την επόμενη εβδομάδα κατά πόσον η νέα επιτροπή θα μας υποστηρίξει από αυτού. Ε, νιώθω κάποιον εκνευρισμό βέβαια, δεν είμαι σίγουρη για την δέσμευση που θα αναλάβει η νέα επιτροπή Κομισιόν. Και πρέπει να τονίσουμε ότι αυτό είναι βασικό και για την οικονομία της Ευρώπης και του κόσμου. Ο υπόλοιπος κόσμος εμάς προσβλέπει. Κάθε φορά που πάω κάπου επίσκεψη μας λένε σε χώρα και μου λένε εσείς φταίτε για τις κλιματικές αλλαγές, τι θα κάνετε λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε κάτι το πολύ στεναρό, ζωτικότατο. Μάλιστα. Έχουμε τώρα πολλούς εγγεγραμμένους ομιλητές πέντε τουλάχιστον. Τρία λεπτά περίπου ο καθένας. Γιατί θα προσθεθούν και άλλοι. Λοιπόν, χέντε χάουταλα. Ευχαριστώ Λίνδα. Δεν είχα το χρόνο να διαβάσω τις σημειώσεις, αλλά θα τις κοιτάξω βέβαια, θα τις κοιτάξω. Θα ήθελα να ζητήσω, να ρωτήσω τους συναδέλφους και εσάς την ίδια, τι θα μπορούσε να γίνει για να απλοποιηθεί η πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών με τη χρησιμοποίηση όλων των αναπτυξιακών μέσων όπως και του Αναπτυξιακού Ταμείου. Διότι πιστεύω ότι εκτός από τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για τη χρηματοδότηση διεθνών μέτρων αντιμετώπισης, πρέπει να βρούμε και καινοτόμους τρόπους να βρούμε νέες λύσεις και δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό το φρονούν και εκείνοι που γράφουν τα προγράμματα δράσης για το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Ταμείο. Αυτό να το δούμε. Ποιοι καινοτόμοι τρόποι μπορούν να βρεθούν. Δεύτερον, από ό,τι έχω παρατηρήσει, η σύμβαση για τα κλιματολογικά σκοντάφτει πάντα στην έλλειψη θέλησης των βιομηχανιών, των αναπτυσσομένων κυρίως χωρών. Με τι τρόπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αναπτυξιακά εργαλεία για να ενθαρρύνουμε και τις χώρες του ΓΑΜΑ 77 ή του ΖΙΤΑ 77, τις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες να αναλάβουν τη δέσμευση να πάρουν τέτοια μέτρα και να εγκριθεί η σχετική συνθήκη. Δεν έχω συγκεκριμένε ιδέες, αλλά θέλω να ζητήσω να τα σκεφτούμε. Γκερέρο. Ευχαριστώ. Όπως είπε και η πρόεδρος Μακάβεν, Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τελικά ποιος είναι ο κίνδυνος για την ανθρωπότητα αν δεν ανταποκριθεί θετικά στις κλιματικές αλλαγές. Στην πραγματικότητα οι κλιματικές ε, αλλαγές έχουν να κάνουν όχι τόσο με το τι είδους μέλλον θα έχουμε, αλλά με το αν θα έχουμε μέλλον. Διότι οι αλλαγές είναι αλυσιδωτές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το υπογραμμίσουμε αυτό, γιατί το να αρνούμεθα ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, δυστυχώς είναι κάτι που ισχύει σε αρκετές χώρες μας και σε αρκετές κυβερνήσεις. Η οικονομική δε κρίση αποτελεί συχνά άλοθη για αυτούς που δεν θέλουν να υιοθετήσουν μέτρα για να καταπολεμήσουν την κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, στην προηγούμενη θητεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε γκρίνει ψήφισμα για την πολιτική όσον αφορά το κλίμα. Η θέση του Κοινοβουλίου λοιπόν ήταν πιο φιλόδοξη από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά δηλαδή τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ή τις ε, δεσμεύσεις που θέλουμε να πάρουμε για διάφορα ζητήματα. Για την ενεργειακή απόδοση για παράδειγμα, όπου εκεί δεν υπήρχε Σαφή πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να, που είχε πει ότι θα υπέβαλε μια πρόταση το φθινόπωρο να μας πει προλαβαίνουμε να πάμε με κάποια περηφάνεια στην διάσκεψη για το κλίμα που θα γίνει στη Λίμα. Προλαβαίνουμε. Θέλω επίση να υπογραμμίσω ότι από πλευράς της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής το βασικό σημείο είναι πώς θα βοηθήσουμε εκείνε τις χώρες, του τομεί τα εδάφη, όπου η κλιματική αλλαγή έχει πιο καταστροφικές συνέπειες. Αναφέρθηκε στην Κένια για παράδειγμα, ε, αυτό δεν ήταν, ναι. Υπάρχουν όμω πολλέ χώρες όπου αποδεικνύεται ξανά και ξανά ότι πιο φτωχοί είναι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από οποιαδήποτε κλιματική αλλαγή. Υποφέρουν και οικονομικά και περιβαλλοντικά. Εμείς λοιπόν πρέπει ως Επιτροπή Ανάπτυξης να δεσμευτούμε με την πολιτική για το κλίμα, να έχουμε και μια πολιτική αλληλεγγύης προς τις χώρες αυτές που από μόνες τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά υφίστανται τις συνέπειες από τη γενική κατάσταση στον κόσμο. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το σχολιάσει αυτό. Βεβαίω, ναι, και μετά από λίγο και στο τέλος. Κύριος Πάγκα και μετά η Καθλίν Φαν Μπρέμπτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, να κάνω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον είναι ζωτικό να επιτευχθεί συμφωνία στα πλαίσια του ΣΚΟΠ ώστε να μειωθεί η εκπομπή αερίων θερμοκηπίου διότι ο πλανήτης μας ζεσταίνεται, θερμαίνεται. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια σαφή θέση για να επιτευχθεί αυτή η διεθνή συμφωνία. Γίνονται προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μειωθούν οι εκπομπές και αυτό θέτει την Ευρώπη στο προσκήνιο για τα κλιματολογικά και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να επηρεάσει θετικά τις διεθνείς αξέλιξους προς αυτό. Δεύτερον, για τις χώρες της Αφρικής που υποφέρουν και αυτές από τις κλιματολογικές αλλαγές, ιδιαίτερα το οι χώρες η τα μικρά νησιά του Ειρηνικού υποφέρουν περισσότερο από όλα και θα χρειαστεί να προσαρμοστούν στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Είναι θέμα αξιοπιστίας της Ένωσης και συνέπειας και συνοχής των προγραμμάτων μας. Ευχαριστώ. Κατρίν Βαν Μπρέντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο. Θέλω μόνο να αναδιατυπώσω αυτά που είπα στη συζήτηση της προηγούμενης εβδομάδας. Εγώ είμαι καινούρια στην Επιτροπή σας και ακόμη μαθαίνω. Ξέρω όμως μερικά για την κλιματολογική πολιτική στην Ευρώπη και θα είμαι και εγώ στην αντιπροσωπεία μας στη Λίμα και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η Επιτροπή ΑΝΑΠΤ γνωμοδοτεί για τις κλιματολογικές αλλαγές. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι έχουμε πολλά χρήματα να δαπανίσουμε αλλά τελικά θα φανεί ότι όλα αυτά δεν έχουν καμιά σημασία σε σύγκριση με τα ποσά που χρειάζονται πράγματι για να σωθεί ο πλανήτης η βιομηχανία και οι οικονομίες μας. Αυτό ήθελα να τονίσω, αλλά το είπατε κι εσείς, Πρόεδρε. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής, ε, την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το σημαντικότερο ως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ότι δική μας ευθύνη είναι και πρέπει να ντρεπόμαστε από αυτά, για αυτά που κάναμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια γιατί δεν αναλάβαμε τις ευθύνες μας. Επίσης μιλήσατε για το ότι χρειάζονται σαφείς στόχοι για την αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών αλλά και για τα ενεργειακά και για την αποδοτικότητα της ενέργειας. Και τα τρία είναι πολύ σημαντικά μαζί και το προσεχές συμβούλιο θα είναι ζωτικό. Θα το λέει και το ψήφισμα μεν, αλλά ήθελα να είμαστε βέβαιοι ότι θα τα ακούσει αυτά και η Επιτροπή Περίφ και τελικά η Ολομέλεια και μετά θα μπορέσουμε να πάμε στη Λίμα. Καλό είναι που υπάρχουν εδώ άνθρωποι από την Περιφερειακή Επιτροπή να τα ακούσουν. Ο κύριος Ρούμπικ. Κοιτάξτε, μια που είμαι από την Επιτροπή Βιομηχανίας, οφείλω να συγχαρώ την κυρία Χέντεγκαρτ για το τοποθέτησε τον στόχο του 20% και τον εφάρμοσε πάρα πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υπόδειγμα παγκοσμίω και εδώ πέρα έχει βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν ε, ε, μειώνουμε τόσο πολύ τις ε, εκπομπές μας. Ε, είμαστε λοιπόν θα έλεγα υπόδειγμα προς αυτό και όταν κάποιοι μιλούν για αποτυχημένη πολιτική στην Ευρώπη αναρωτιέμαι τι πρέπει να πει ο υπόλοιπο πλανήτης δηλαδή εδώ πέρα. Το σύστημα εμπορίας εκπομπών πρέπει να το ξανασκεφτούμε να μην οδηγήσει στο να φύγουν οι βιομηχανίε μα από εδώ και να πάνε να παράγουν αλλού με χειρότερες συνθήκες και με χειρότερο αποτέλεσμα τελικά για το κλίμα. Εξάλλου και η αγοραστική μας ε, δύναμη ωφελείται όταν παράγουμε, όχι όταν εισάγουμε. Οπότε καλό είναι στα εισαγόμενα προϊόντα να δούμε έναν δείκτη διοξιδίου του άνθρακα για να ξέρουμε ότι στη χύψη χώρα ή στο χύψη προϊόν ε, υπάρχει αυτή η εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα για να μπορεί και ο καταναλωτής να κάνει κάτι για να μειώσει τις εκπομπές. Αυτό ειδικά εν ώψη της διάσκεψης των μερών είναι μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση. Πώς θα έχουμε ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κοράλ και μετά Λόλα Σάντσες. Ε, ευχαριστώ. Εγώ μελέτησα το κείμενο αυτό Αλλά αυτό που θέλω να πω για την κλιματική αλλαγή είναι ότι οι επιπτώσεις δεν μπορεί να συνεχίζονται για τον πολίτη, για τον πλανήτη μας, συγγνώμη. Το 2015 στο Παρίσι θα αποφασίσουμε για την περίοδο μετά το Κιώτο. Αλλά λίγο πολύ έχει αποφασιστεί να μην αποφασίσουμε. Γιατί... Και τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι αναβάλουμε τις δράσεις για αργότερα, για το 2020 και μετά. Αλλά εγώ θέλω εδώ να επανέλθω σε δύο ζητήματα όσον αφορά το πράσινο ταμείο για το κλίμα και τα μέτρα αποζημίωσης. Όσον αφορά λοιπόν αυτό το πράσινο ταμείο που συζητήθηκε το 2010 στο Κανκούν έχει να κάνει με τις υπονάπτυξη χώρες που απειλούνται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Αλλά από ό,τι φαίνεται το ταμείο αυτό έχει κάποιο είδους διπλωματική ασυλία και δεν θα μπορεί να ελεγχθεί ούτε ποινικά ούτε αστικά από τις δικαιούχες χώρες. Πρόκειται όμως για πολύ σημαντικά ποσά, 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχουμε συνεπώς την αίσθηση ότι κάπου κρύβεται διαφθορά εδώ. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν, πιστεύω εγώ, να διαχειριζόμαστε το ταμείο αυτό με απόλυτη διαφήνεια. Ε, διαφάνεια. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα αντιστάθμισης, ξέρουμε ότι υπάρχουν μηχανισμοί ανάπτυξης για να μειωθούν οι εκπομπές σε τρίτες χώρες που υφίστανται κλιματικές αλλαγές από άλλες χώρες που ρηπαίνουν. Αυτό βέβαια έχει σημαντική συνέπεια πάνω στους ντόπιου ε, έχουν μελετηθεί κάποιοι μηχανισμοί και θα μπορούσαν να υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στους κατοίκους τρίτων χωρών. Η κυρία Σάντσεθ. Ευχαριστώ. Έχω διάφορα σχόλια σύντομα. Θέλουμε το κόστος να το αναλάβουν οι αναπτυγμένες χώρες γιατί ιστορικά έχουν ευθύνη, γιατί έχουν ένα περιβαλλοντικό χρέος συσσωρευμένο πολλά χρόνια. Και επίσης προτείνουμε, αν και εμφανίζεται στο σημείο 5 κάπως, και έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, αλλά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται αυτό παράλληλα Υπάρχουν επιπλέον κονδύλια δηλαδή από την ανάπτυξη. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξει τη θέση αυτή και σε άλλα φόρα όπως είναι ο ΙΕ ή ο ΣΑ. Να μην μπερδεύονται δηλαδή τα κονδύλια, να πρόκειται για ένα νέο κονδύλιο χωριστό. Ευχαριστούμε Γκέρενς και μετά η κυρία Χολμπρουκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο σημεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Το ένα έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση και το άλλο έχει να κάνει με τη συνοχή της πολιτικής μας. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, βλέπω στο σχέδιο ψηφίσματος, στο σημείο... Μόλις το είχα δει. Στο Δέλτα, μάλλον, που αναφέρονται 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2020. Με την εμπειρία που έχουμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση, μας χρειάζονται πολύ περισσότερα. Πολύ εδώ στην Επιτροπή αυτή έχουμε υπενθυμίσει ότι όχι ό,τι έχει να κάνει με την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής ε, αλλαγής πρέπει να χρηματοδοτούνται από άλλο κονδύλι, επιπλέον από την ανάπτυξη δηλαδή, και όχι μέσα από την ανάπτυξη. Ομόφωνα συμφωνήσαμε σε αυτό το σημείο. Και οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως πάντα ξεφεύγανε για αυτό το θέμα. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να βρούμε τα 8 δισεκατομμύρια στην Κοπεχάγη, Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη. Γι' αυτό είναι ψευδέστηση ή λέμε συλλογικά ψέματα αν λέμε ότι θα έχουμε τα χρήματα αυτά για το 2020. Εγώ πολύ θα ήθελα, αλλά δεν το βλέπω. Εξού, ανάμεσα στο όλα ή τίποτα, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές και να επιμείνουμε στην συνοχή της πολιτικής μας. Αφήνουμε μόνη της τη Γερμανία με την ενεργειακή της επανάσταση να μας δείξει το δρόμο. Μα αν μία χώρα αποτύχει, τι θα γίνει, θα αποτύχουμε όλοι. Και αν μία πετύχει, θα πετύχουμε όλοι. Συνεπώς πρέπει να πετύχει. Σε θέματα λοιπόν μείωσης αερίων του θερμοκηπίου, αυτά τα δύο στοιχεία πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι διακινδυνεύουμε να απογοητεύσουμε για άλλη μια φορά τις υποανάπτυξη χώρες με ποσά τα οποία δεν θα μπορέσουμε να βρούμε ενώ θα βρούμε ένα περιλάχιστο ποσό σε σχέση με τα 100 δις που χρειάζονται. Η κυρία Χόλμπουκ, τελευταία. Μίλησαν πολύ για λεφτά, για κατανομή του κόστους. Πρέπει να δούμε τα πρακτικά, πώς θα εξασφαλίσουμε τη διατροφική ασφάλεια, γιατί ειδικά δεδομένης κλιματικής αλλαγής οι γεωργικές επιχειρήσεις και τα γεωργικά μοντέλα στις ε, περιοχές ε, οι οποίες ε, πλήττονται πιέζονται πάρα πολύ. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να μοιράσουμε λεφτά, αλλά πρακτικά πράγματα που πρέπει να λυθούν. Μοντέλα γεωργίας που θα ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή και θα μπορούν να σταθούν. Γιατί μόνο έτσι θα διασφαλιστεί το δικαίωμα στη διατροφή. Υπάρχει ανθρώπινο δικαίωμα στην διατροφή, αλλά δισεκατομμύρια άνθρωποι πεινάνε. Οπότε θα είναι μεγάλη η πρόκληση και πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Είναι σχέδιο αυτό, θα πάει στη μετάφραση, θα λάβετε τη μετάφραση σε δύο εβδομάδες και μετά μπορείτε να κάνετε τροπολογίες. Πριν πάμε παρακάτω, εγώ θα ήθελα να ακούσω τι έχει να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα έχουμε και σύνοδο κορυφή στη Νέα Υόρκη. Νομίζω είναι εκεί ο πρόεδρος Μπαρόζο. Δεν ξέρω τι θα πει. Πείτε μας εσείς. Και να απαντήσετε σε κάποιε ερωτήσεις. Άντλμπερτ Γιάννη από τη Γενική Διεύθυνση Κλίματος. ξεκινήσω ευχαριστώντας ε, το Κοινοβούλιο για τον ενδιαφέρον του ειδικά την Επιτροπή ΔΕΒΕ. Οι διαπραγματεύσεις, όπως είπε η κυρία Μακάβανς, πραγματικά είναι σε κρίσιμη φάση φέτος. Όπως ξέρετε, η Σύνοδος Κορυφής του Μπανκιμούν λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Επιπλέον, και η διάσκεψη της Λίμας ε, θα είναι σημαντική. και ελπίζουμε να έχουμε μια νέα παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Είμαστε λοιπόν σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο που έχει αλλάξει από την Κομεχάγη και δόθε και μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Βλέπουμε πραγματικά πως οι βασικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνουν εσωτερικά μέτρα περισσότερα από ό,τι στο παρελθόν, ειδικά αν δει κανείς της ΕΠΑ και την Κίνα, όπου έχουμε άνευ μέτρα άνευ προηγουμένου. Εκεί πέρα υπάρχει ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών που ακολουθεί, θα έλεγα, το παράδειγμα της Ένωσης. Και, κοιτάζοντας και το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι προφανές πως η επιτυχία της Ένωσης να συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη και τη μείωση των εκπομπών είναι κάτι το οποίο πλέον αναγνωρίζεται Πρέπει επίσης να συνεχίσουμε στην πορεία αυτή και όπως ίσως ακούσατε, σύμφωνα με την ε, έκθεση του διακυβερνητικού πάνελ, αν δεν έχουμε μια σωστή συμφωνία στο Παρίσι, πάμε προς έναν κόσμο με αύξηση θερμοκρασίας 3,5 με 4 βαθμούς μέχρι το τέλος του αιώνα, που θα επηρεάσει πολλούς τομείς και στην Ευρώπη και το βιός των ανθρώπων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό ενδιαφέρει την Επιτροπή σας. Ε, πρέπει να θυμόμαστε πως η κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση όσον αφορά την ανάπτυξη. Οι χώρες με τις μεγαλύτερες ανάγκες είναι και πιο ευάλωτες. Και ταυτόχρονα όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν την πρόκληση του να αναπτυχθούν ε, με έναν τρόπο συμβατό ε, με την μείωση της κλιματικής αλλαγής. Εάν λοιπόν η αναπτυξιακή βοήθεια δεν συνεισφέρει σε αυτό το στόχο, θα υπονομεύσει τους στόχους της. Οπότε, κατά την απόψή μας, οι ανθρώπινοι στόχοι της ανάπτυξης και οι κλιματικοί στόχοι ε, πραγματικά πάνε χέρι-χέρι. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάσκεψη της Λίμας. Πρώτα απ' όλα, να ξέρει το τι γίνεται όσον αφορά τις ε, πληροφορίες ε, που θα υπάρχουν εκ των προτέρων ένα τεχνικό ζήτημα καθώς πέρσι στη Βαρσοβία όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να έχουν κάποια σχέδια δεσμεύσεων για τις εθνικές συνεισφορές στην μείωση των εκπομπών πολύ πριν από την διάσκεψη των Παρισίων και το να συμφωνήσουμε επί των ζητημάτων αυτών σημαίνει πως θα ε, συμφωνήσουμε στις ε, συνεισφορές με τρόπο συγκρίσιμο και κατανοητό. Γιατί έτσι ελπίζουμε να έχουμε και μια διεθνή διαδικασία που θα μας επιτρέψει πριν, από, πριν πάμε στο Παρίσι να ξέρουμε εάν είναι επαρκείς αλλά και δίκαιες αυτές οι ε, συνεισφορές. Ε, το άλλο πράγμα το οποίο έχουμε ως στόχο είναι περαιτέρω πρόοδος ε, στο πώς η νέα αυτή συμφωνία μπορεί να δει το ζήτημα της χρηματοδότησης της προσαρμογής. Και ακριβώς στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αξιόπιστη όπως είπατε. Αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα από τον πρόεδρο Μπαρόζο είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στείλει 14 δισεκατομμύρια σε εταίρους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα επόμενα 7 χρόνια στο πολιετές πρόγραμμα και πρέπει και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες να συνεισφέρουν. Και οι αναπτυσσόμενες επίσης ε, θα συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση αυτή και επίσης να φροντίσουμε η συμφωνία αυτή να αντιμετωπίζει το ζήτημα της ιδιωτικής χρηματοδότησης, καθώς, όπως είπε η κυρία Μπέρντερ, ε, η πρόκληση είναι τέτοια ώστε δεν επαρκεί η δημόσια χρηματοδότηση. Επίσης, ε, τέθη το ζήτημα του τι προσφορά θα κάνει αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Λίμα και πέρα από τη Λίμα όσον αφορά τις δικές μας μειώσεις. Και στο πλαίσιο αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ σημαντικό ε, να παίξουμε έναν ηγετικό ρόλο. Ο κόσμος προσβλέπει σε εμάς. Ε, να έχουμε μια φιλόδοξη πρόταση και αναμένουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 Οκτωβρίου. Οπωσδήποτε θα γίνει κάτι πριν πάμε στο διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ και θα το υπενθυμίσει άλλωστε και ο πρόεδρος Μπαρόζο σήμερα. Και μετά, τέλος, όσον αφορά το τι θα γίνει πριν από το 2020 σε άλλα πλαίσια που αφορούν τα κίνητρα για άλλες δράσεις για πολλούς ενδιαφερόμενους πράγματι για να απαντήσω τον κύριο Κοράο. Οπότε, η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λίμα είναι σημαντική για να πετύχουμε τις προθεσμίες μας και αυτός είναι άλλος ένας λόγος για τον οποίο συμφωνούμε με το, το Κοινοβούλιο θέλει να κάνει μια έτσι, έντονη δήλωση πριν από τη άσκηση της Λίμας. Μάλιστα. 14 Οκτωβρίου η προθεσμία τροπολογιών. Ωραία. Τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ. Περνάμε σημείο 8. Ψηφοφορία για το Γενικό Προϋπολογισμό για το 15 Είναι, αφορά τη γνωμοδότηση. Ψηφίσαμε τις τροπολογίες στην προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής κύριος Ρούμπικ θέλει να πει τίποτα ή αν μπορούμε κατευθείαν να ψηφίσουμε κατευθείαν. Υπάρχει μια συμβιβαστική ψηφοφορία από το ΕΛΚ, σοσιαλιστές και φιλελεύθερους για τις τροπολογίες 2, 3 και 4. Και το έχετε στον κατάλογο. Ναι, το έχετε. Ξέρω ότι έχετε και μια προφορική τροπολογία, άλλο αυτό. Στο τέλος του τυπωμένου καταλόγου είναι οι συμβιβαστικές, οι συμβιβαστικοί. Πριν αρχίσουμε λοιπόν, θα δοκιμάσουμε το μηχάνημα γιατί προηγουμένως είχε πρόβλημα. Εικονική ψηφοφορία λοιπόν ποιος είναι υπέρ ενός καφέ. Άρχεται η ψηφοφορία. Έλξε. Η ψηφοφορία είναι υπέρ του καφέ ή του τεΐου. Δεν θα μας φέρουν βέβαια, αλλά τέλος πάντων απλώς δοκιμάζαμε. Εγώ δεν μπορώ ούτε καφέ ούτε τσάι γιατί δεν έφερα την κάρτα μου. Μπορείτε λοιπόν να λαμβάνετε υπόψη την ψήφο μου κάθε φορά. Ναι, θα μας λέτε κάθε φορά ναι ή όχι. Αν χρειαστεί με κάρτες ψηφοφορία. Αν. Λοιπόν... Άλλος χωρίς κάρτα. Δεν δουλεύει, ε, αλλάξτε θέση. Πολλοί δεν έφεραν, αν πολλοί δεν έφεραν κάρτα θα, γίνουν, θα δυσκολέψουν τα πράγματα. Λοιπόν, έχει όλο ο κόσμος την κάρτα του, δουλεύουν οι κάρτες. Κυρία Σλάιν δουλεύει, καλά. Αν δεν δουλεύει να μου το πείτε. Αρχίζουμε λοιπόν την αληθινή ψηφοφορία. Προφορική τροπολογία στην 1. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, να σας διαβάσω. Λέει, καλούμε, ζητούμε αύξηση της χρηματοδότησης των ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως την υπάτη αρμοστία, τους, ε, τους χωρίς σύνορα κλπ. Ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση των κρίσεων στο, Σιράκ, στο Ιράκ, Συρία και Γάζα για να μπορέσουν οι πρόσφυγες εκεί να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες, ιατρική περίθαλψη και αντιμετώπιση του ιού έμπολα. Είναι λοιπόν τροπολογία που αντικαθιστά τη χωριστή την κατατμήματα ψηφοφορία που προβλέπει ο κατάλογος. Δέχεστε όλη την προφορική τροπολογία μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ή μάλλον όχι, διαχειρός ε, η ανατάσεως υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά χες εγκρίνεται. Τροπολογία 2 η... Α, όχι, καταπίπτει, καταπίπτουν όλες αυτές. Πάμε στην 5 για την παράγραφο 6. Α, έχει αποσυρθεί, έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 6. 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, καταπίπτει. Ή δηλαδή απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 του κυρίου Ρούμπικ. Υπέρ, Κατά. Εσ. Εγκρίνεται. Οκτώ. Α, όχι, αφού λέει καλύπτεται. Και ε, πρέπει να μου το πείτε. Καλύπτεται. Δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε λοιπόν. Τη γνωμοδότηση ο σύνολό τη είπε Τα. εγκρίνεται αλλά τώρα ηλεκτρονικά. Ε, ηλεκτρονικά έπρεπε μου λένε για το σύνολο. Άρχεται η ψηφοφορία. Συν μία ψήφο υπέρ της κυρίας Χάλταλα Ελξέι 24 υπέρ 3 κατά εγκρίνεται η νομοδότηση. Ευχαριστώ. 9 διάφορα. Έχει κανεί τίποτε να θέσει στα διάφορα. Ορίστε κυρία Χαοταλά μου. Αφού έχουμε λίγη ώρα. Είχα ξεχάσει στους συντονιστές να μιλήσω για την επιστολή που έστειλαν 46 ευρωβουλευτές στο Γιούνκερ λέγοντας ότι θέλουν αλλαγές στη σύνθεση της Κομισιόν και στις δικαιοδοσίες αρμοδιότητες των επιτρόπων, μεταξύ των οποίων και για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα μέλη της Επιτροπής μας και εσείς η Ιδία, μήπως μπορείτε να διασφαλίσετε τι θα γίνει με αυτό γιατί είναι παλαιομοδίτικη μέθοδος αυτή και είναι απαρχαιωμένο το ότι δεν προβλέπεται καθόλου τέτοια αρμοδιότητα στη Νέα Επιτροπή. Δεν το έχουν συζητήσει οι συντονιστές, θα το συζητήσουν μετά οι ομάδες και ύστερα θα φανεί από ερωτήσεις στις ακροάσεις. γιατί δεν θα προλάβουμε μέχρι τους επόμενους συντονιστές. Ο κύριος Γκέρνης. Δεν αντέδρασα προηγουμένως γιατί δεν πρόλαβα σε αυτά που είπε για τις κλιματολογικές αλλαγές ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Προηγουμένως είχα επιμείνει ότι τα χρήματα που χρειάζονται για την καταπολέμηση των αποτελεσμάτων των κλιματολογικών αλλαγών στις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με βάση έναν προπολογισμό διαφορετικό από τον αναπτυξιακό. Ενώ η Κομισιόν είπε ότι αν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα αναπτυξιακά χρήματα τότε δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Ενώ εγώ θεωρώ ότι αν θέλουμε να πάρουμε λεφτά από την ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές τότε δεν καταλήγουμε πουθενά. Γιατί εμάς η απόφασή μας ήταν αυτή ακριβώς που σας είχα πει. Είπα ακριβώς αυτά που είχαμε συμφωνήσει στην προηγούμενη θητεία και θα ήθελα να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη της επόμενης μας συνεδρίασης. Ε, προτείνεται το στους συντονιστές και θα δούμε. Ωραία. Δεν υπάρχουν διάφορα. Σας είπα για τις ακροάσεις της επόμενη εβδομάδα και την ψηφοφορία για το βραβείο Σάχαροφ. Τώρα θα πάμε στην αίθουσα 2Q2 για την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων Σάχαροφ. Ευχαριστώ για τη σημερινή σας προσέλευση και θα σας δω τη Δευτέρα για τις ακροάσεις.